Ε, στρέψουμε το βλέμμα στο αύριο και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, απόλυτα την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κοράτσα Βίλντα. Συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία για την ε, έκθεση της συναδέλφου Κοράτσα Μπίλ θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που αφορά στην έκθεση της κυρίας Λεγκρίπ για τον ενωσιακό τελωνιακό κώδικα και θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτρια να πάρει πρώτα το λόγο για τέσσερα λεπτά. Madame Le Grip. Merci, Madame euh, la Présidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Απόψε εδώ συζητάμε το κείμενο της έκθεσής μου για τον τελωνιακό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κείμενο το οποίο, στο οποίο καταλήξαμε μετά τον τριμερή διάλογο με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και με την παρουσία του Συμβουλίου από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο του 2013. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της διαπραγματευτικής ομάδος, ιδίω τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, τον πρόεδρο Μάλκον Χάρμπορ που ήταν βράχος της διαπραγματεύσης, όπως επίσης και τις υπηρεσίες υπηρεσίε του Κοινοβουλίου, την Γενική Διεύθυνση Ταξού, την Προεδρία την, του Συμβουλίου, που όλε οι Προεδρίε κατέβαλαν ιδιαίτερε προσπάθειε και όλοι μαζί κατορθώσαμε να φτάσουμε σε συνένεση και πιστεύω ότι η ψηφοφορία που έγινε στις 29 Μαΐου ε, επιβεβαίωσε την επιτυχία των εργασιών μας. Η Τελωνιακή Ένωση έχει κεφαλαιόδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1957, από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης υπάρχει και αποτελεί ένα πυλώνα στον οποίο βασίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και βάσει αυτού λειτουργούν σημαντικές κοινοτικέ πολιτικές και η υπηρεσία τους και η αποτελεσματικότητά τους ε, αποτελούν ε, μέλημα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έκθεση αυτή ε, που θα ψηφιστεί αύριο ε, προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε ε, τον τελωνιακό κώδικα. Αυτός ο τελωνιακός κώδικας που ισχύει τώρα υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και σκεφτείτε τα, τις τεράστιες αλλαγές που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια. Παγκοσμιοποίηση, εντατικοποίηση των εμπορικών σχέσεων, τεχνολογικές και τεχνικές πρόοδοι σημαντικές εξελίξεις και νέες προκλήσεις. Είτε αυτό είναι τεχνολογική κίνδυνη, είτε είναι κίνδυνη τρομοκρατίας, είτε είναι υγειονομική κίνδυνη, είτε πρόκειται για την εξέλιξη της απομίμησης και του λαθρεμπορίου και αναφέρω μόνο λίγους από αυτούς τους τομείς εξελίξεων. Εξυγχρονισμός λοιπόν και ευελιξία είναι αυτά τα οποία χρειάζονται σε αυτή τη μεταρρύθμιση της τελωνιακής νομοθεσίας που θέλουμε να επιτύχουμε, δημιουργώντας ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις και διαφορετική μεταχείριση στα κράτη-μέλη και αυτό θέλουμε να το συνδυάσουμε με την αποτελεσματικότητα και τις απαιτήσει που έχουμε στον τελωνιακό τομέα. Θα αναφέρω μόνο τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις ε, που προσπαθούμε να επιφέρουμε στο κείμενο. Θέλουμε να έχουμε τελωνία χωρίς ε, έντυπα, αλλά μόνο με ηλεκτρονική με ηλεκτρονική διακίνηση. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ε, να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, να έχουν ένα πιο εύκολο περιβάλλον στην επιχειρηματική του δραστηριότητα και στις συναλλαγές τους με τα τελωνία. Θα δώσουμε εργαλεία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να συνεργαστούν καλύτερα με τις επιχειρήσεις εταίρους τους σε ολόκληρο τον κόσμο κυρίως μέσω του μηχανισμού αμοιβαίας αναγνώρισης. Και θέλω να προσθέσω στον κατάλογο των σημαντικών εξελίξεων, ε, την μεταρρύθμιση της προσωρινής αποθήκευσης εμπορευμάτων για να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα εργαλεία μας και πρέπει να προχωρήσουμε με βάση αυτά τα εργαλεία. Η διαδικασία μεταρρύθμισης από το 2008 έχει ε, αντιμετωπίσει προβλήματα και με την οικονομική κρίση έχουν δημιουργηθεί ακόμη περισσότερα προβλήματα. Τώρα πλησιάζουμε σιγά σιγά στο στόχο μας και θέλουμε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο μεταρρυθμίζει την ε, Τελωνιακή Ένωση και χρειάζεται ε, όλη η προσπάθεια που μπορούμε να καταβάλουμε για να μπορέσουμε αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε σκόπιμα να εφαρμόσουμε μαζί με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Θέλουμε να δώσουμε στην εσωτερική αγορά και σε όλου του φορεί τη εσωτερική αγορά ε, όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση. Εφόσον μπορούμε να υποφεληθούμε, θα μα δώσει ε, πολλά καλά στοιχεία. Θέλουμε να εγγυόμαστε το υψηλό επίπεδο προστασία τη εσωτερική αγορά ε, και των καταναλωτών μα, ενώ παράλληλα θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει στον 21ο αιώνα με όλο τη το δυναμικό. Αν μου επιτρέπετε πρόεδρε θέλω να τονίσω κάποια θέματα. Η υλοποίηση του κώδικα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι εξίσου σημαντική όπως και η αυριανή ψηφοφορία και όλη η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Θέλουμε να δώσουμε στην Επιτροπή και στις τελωνιακές υπηρεσίες ένα εργαλείο για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν όλα αυτά είναι θεμελιώδου σημασία κατά την προετοιμασία όλων των τεχνικών διατάξεων και όλων των συγκεκριμένων και πρακτικών λεπτομεριών πίσω από τι οποίες καμιά φορά κρύβονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, θέλουμε να συνενώσουμε όλους τους εμπλεκομένους, όλους τους ενδιαφερομένους, ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια, ώστε από τον διάλογο και από τη συζήτηση να καταλήξουμε στο τέλειο αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι οδηγίες που σίγουρα έχετε δώσει στις υπηρεσίες σα, κύριε Επίτροπε και σίγουρα αυτό θα είναι το πνεύμα στο οποίο θα δουλέψουμε στο μέλλον και όλοι θα συνεργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Λεγκρίπ, επίτροπε Σεμέτα, καλώ ορίσατε για το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Σίγητρια, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Ο νέο κανονισμό για τον τελωνικό κώδικα, τον οποίο σήμερα συζητούμε, αποτελεί ένα παράδειγμα του πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις. Κυρίως πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Χάρμπορ και κυρία Λεγκρίπ για όσο πετύχανε, για το πόσο αποφασιστική ήταν, ούτως ώστε να τηρήσουμε και τους στόχους, αλλά και το χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τον τελειωνιακό κώδικα. Πολύ θεωρούσαν ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Όλα αυτά γίνανε σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Επίση, αντιμετωπίστηκαν ένα σωρό δυσκολίε. Και έτσι και τα τρία θεσμικά όργανα ικανοποιήθηκαν. Προσωρινή αποθήκευση και οι Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο από ό,τι είχαμε προηγουμένως. Τώρα θέλω να σας τονίσω τρεις θεμελιώδεις αρχές που πολύ συχνά τις ξεχνούμε. Πρώτα πρώτα, η ασφαλεία δικαίου που μας παρέχεται από αυτούς τους νέους κοινού κανόνες. Έτσι θα έχουμε ενιαία εφαρμογή του ενωσιακού τελωνικού κώδικα θα εξορροπήσουν την αξιοπιστή που να υπάρχει πλευρά αλλά και την ε, συνέπεια εφαρμογή τη νομοθεσία. Επίση, έχουμε τώρα το νέο περιβάλλον χωρί έντυπα. Αυτό αντιστοιχεί στην ε, σημερινή κατάσταση κατά την οποία θέλουμε να έχουμε μια όμορφη εφαρμογή, αλλά χωρί ε, πολλά χαρτιά, χωρί χαρτοβασίλειο. Επομένω, έτσι νομίζουμε ότι θα εξοικονομηθεί πάρα πολύ χρόνο υπέρ του εμπορίου. Επίση, να δούμε τώρα πώ θα έχουμε την επιβεβαίωση μεταξύ των, των, ε, των τελωνίων και των ε, ε, νομίμως συναλλασσομένων εμπόρων. Αυτό έχει να κάνει επίση με του ε, ε, νόμιμους συντελεστέ του εμπορίου και είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε συμφωνήσει, αλλά σήμερα για την προηγούμενη σου νομοθεσία αυτό δεν είχε ρυθμιστεί ρητά. Τώρα πάντως έχουμε μια πάρα πολύ στιβαρή νομική βάση ούτως ώστε να μπορέσουμε να θεσμοθερήσουμε το υπήν την σχέση αυτή τελωνίων θεσμών οργάνων για το μέλλον και επίση έτσι μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε από την βασική νομοθετική πράξη προς την εφαρμογή. Σήμερα δεν θα πρέπει να σας διαβιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επίτροπη πρόκειται να τηρήσει και να συνεχίσει την πορεία από τις προβοσιακές εργασίες προς τις μέλουσες κατανάθεση κατουσιώδης πράξεις. Επίσης έχουμε κάποιους ειδικού, έχουμε κάνει μια προπαρασκευή με κάποιο είδου ε, διάφανη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμπορίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτέλους το Κοινοβούλιο ψηφίζει μια έκθεση που θα δικήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που υπάρχουν στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Ανισότητες που είχαν αρνητικές επιπτώσεις και στους καταναλωτές, όχι μόνο στους υπεύθυνους. Πολλές φορές τονίσαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία ενιαία αγορά, μία σωστή αγορά, αν υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες στα σύνορα, διαφορετικά, διαφορετικά ωράρια λειτουργίας, ε, άτομα που είναι διακριμένα, ε, επισήμως και ανεπισήμως, και καθώς και διάφορα ποσοστά ΦΠΑ. Αυτές είναι διαφορές που χωρίζουν τους μεγάλους του Βορρά και υπάρχει πολύ μεγαλύτερος έργος και για όλα αυτά ε, εντείνουν ε, τι ανισότητες θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί και οι ίδιοι κανόνε. Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά η οποία να εγγυάται την, ε, κάτι στου καταναλωτέ όσο οι ευρωπαϊκέ χώρε ε, δεν κάνουν ενιαίο το τελωνιακό σύστημα. Ελπίζουμε ότι η διαδικασία αυτή να είναι γοργή και να μπορέσουμε να ε, οδηγηθούμε σε μια ανάπτυξη θα πρέπει, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, να ξεκινήσουμε με τον εσυγχρονισμό του τελωνιακού κώδικα. Πολιτικών ομάδων και πρώτα δίνω το λόγο στη συνάδελφο σλοβιεσκα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το, η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την Τελωνιακή Ένωση. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μέσο για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της εσωτερική αγοράς. Η έκθεση του Κοινοβουλίου υπογραμμίζει το στόχο απλοποίηση και δημιουργία καλύτερων συνθήκων για τους επιχειρηματίες. Η Τελωνιακή Ένωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς και μόνον η ενιαίος χαρακτήρας θα μας επιτρέψει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο το δυναμικό του. Η έκθεση αναφέρεται σε μια ενιαία εφαρμογή σε όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει κατά συνέπεια να εκμεταλλευτούν την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων προσώπων του τελωνίου, να αποφύγουν τις επικαλύψεις και διαδικασίες που θα μπορούσαν να αποβούν κατά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η εγκατάλειψη αυτής της αρχής θα μπορέσει να είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές καταστάσεις. Κατά την άποψή μου πρόκειται για μια υγιή αρχή. Κύριε Λεγκρίπη, αναφέρεται σε ένα σύστημα στο οποίο ο επιχειρηματίας θα πρέπει να, μεταβιβάζει τις, να διαβιβάζει τις πληροφορίες μόνο μία φορά. Καλό είναι αυτό με τα νέα συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και θα επιδοθεί η δυνατότητα για έναν ενιαίο έλεγχο. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά την ανανέωση της, του σημείου που αφορά τον εγκεκριμένο ε, οικονομικό φορέα που μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ε, απλοποιήσεις που έχουν γίνει. Με λίγα λόγια, η έκθεση ασχολήθηκε όχι μόνο με τη Λισαβόνα και τον εξυγχρονισμό των διατάξεων στο τελωνίο, στα τελωνία, αλλά θεώρησε την Τελωνιακή Ένωση ω ένα εργαλείο που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα τη εσωτερική Αγορά. Η απλοποίηση για τις επιχειρήσεις και του επιχειρηματίες θα έχει θετικέ επιπτώσει για την οικονομική εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι μια πολύ καλή στιγμή για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αυτή η συζήτηση που γίνεται για τον εξυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα. εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά όλοι αλλά ιδιαίτερα σκληρά εργάστηκαν η κυρία le που μας έδωσε ένα εξαιρετικό κείμενο βάσης και κυρίως ο πρόεδρος της επιτροπής imco ο κύριος harbour ο οποίος διεύθυνε με εξαιρετική μαεστρία τον τρίλογο που κατέληξε σε αυτό το εξαιρετικά ισορροπημένο νομοθέτημα από το οποίο ωφελούνται οι πολίτες της ευρώπης. έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουν οι πολίτες της ευρώπης ότι αυτό το νομοθέτημα το πάρα πολύ τεχνικό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τους ίδιους με αυτό το νομοθέτημα ευνοούνται οι επιχειρήσεις και μάλιστα σε μια εποχή κρίσης σε μια εποχή που πρέπει να τις προωθήσουμε και να τις προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. σε αυτή την ίδια εποχή κρίσης με αυτό το νομοθέτημα ευνοούνται οι πολίτες ιδιαίτερα τώρα που η διακίνηση επικίνδυνων υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί με αυτό το νομοθέτημα επίσης εξασφαλίσαμε ότι δεν υπάρχουν ανισότητες. τα κράτη τα οποία έχουν πρόβλημα με τους πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων μπορούν να πάρουν το χρόνο τους για να προσαρμοστούν αλλά και εκείνα τα κράτη τα οποία ήδη έχουν προοδεύσει μπορούν να συνεχίσουν το δρόμο τους και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές καλά δεδομένα τα οποία να μπορούν να μιμηθούν τα υπόλοιπα κράτη. νομίζω ότι πραγματικά είναι μια εξαιρετική στιγμή για το κοινοβούλιο και θα βοηθήσει αυτό που λέμε και αυτό που όλοι πιστεύουμε ότι χρειάζεται την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς. ευχαριστώ. Έχει δίκιο η κυρία Ράπτη, η κυρία Μποσκαντίνη. Φαίνεται ένα τεχνικό ντοσιά, θα μπορούσε να αποφέρει πάρα πολλά στις, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ε, το ντογκάνα προέρχεται από το Διουάνα, Διβάνι. Ήταν ο χώρος ε, που υπήρχαν πάγκοι όπου μπορούσε κανείς να καθίσει. Το ντογκάνα, το τελωνίο, είχε ταυτιστεί πάντοτε με την αναμονή και συνεχίζει να αποτελεί ένα παράγοντα κόστους ε, για τις επιχειρήσεις. Οι χρόνοι εκτελωνισμού δεν είναι ποτέ ξεκάθαρη. Αυτό συνεπάγεται κόστος και Συνεπώ κόστος, συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πόρους και χρόνο, εβδομάδες ολόκληρες ε, για να μπορέσουν οι ιδιώτες, ε, οι επιχειρηματίες ε, να μπορέσουν να βγάλουν ένα στεναγμό ανακούφισης. Επιτέλους εκτελονίστηκε το εμπόρευμα. Ο Τελωνιακό κώδικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική εργασία που κάνει το Κοινοβούλιο και μέσω του τριλόγου το, η προσπάθεια που κάνει να στηρίξει αυτό το νομοθέτημα σε συγκεκριμένες προτάσεις. Τονίζει το θέμα της, ε, ε, των τεχνολογιών και της πληροφορικής. Αυτό επιτρέπει ε, εξοικονόμηση και απλότητα. Επίσης αναφέρεται σε ένα ενιαίο σύστημα και μόνο περιστασιακές και για συγκεκριμένους λόγους εξαιρέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει ένα και μοναδικό σύστημα για τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά Όπω όπως είπε πολύ σωστά η συγγήτρια, θα αρχίσουμε να έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των χωρών που προηγούνται και των άλλων που έπονται. Θα ε, αυξηθεί το χάσμα. Ε, ε, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση των αποφάσεων πριν από την απελευθέρωση των εμπορευμάτων. Βεβαίω να υπάρχει δυνατότητα και από πλευρά των τελωνίων να έχουν πρόσβαση στα εμπορεύματα γενικέ γραμμέ, οι τροποποιήσει που προβάλλονται από το Κοινοβούλιο είναι αναγκαίε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διαρευνηθεί η ιδέα που προτάθηκε από την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, μια κοινή task force που θα επιτρέψει να ξεκινήσει, να επιτύχουμε το στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τελωνιακή κοινή αρχή για όλε τι χώρε. Έχουμε μια εσωτερική αγορά. Οι χώρε που έχουν σύνορα με τρίτε χώρε έχουν σύνορα που είναι τα ίδια και που έχουν τις ίδιες δεσμεύσεις, τις ίδιες τους ίδιους περιορισμούς για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν ένα επίτευγμα που δείχνει ότι η περισσότερη Ευρώπη θα αποβεί προς όφελος των πολιτών. Να ξεκινήσουμε όμως με τον κώδικα. E η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να διέπεται από μια συνεπή και ενιαία νομοθεσία. Και βεβαίω η ελληνική νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια, πρέπει να υπάρχει εξυγχρονισμό και έτσι θα πρέπει να έχουμε περισσότερο ανταγωνιστικότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι φανδόν υπέρ του να προσδευτεί η τουρκική νομοθεσία και έτσι να μην έχουμε επικαλύψει όσον αφορά τι ε, εμποροοικονομικέ συναλλαγέ. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα μειώσει το κόστο για τι συναλλαγέ και αυτό επίση θα βοηθήσει όσον αφορά τη συμπίεση των ε, τιμών των εμπορευμάτων και το υπέρ των καταναλωτών και βέβαια αυτό ε, βοηθά τους οικονομικούς ε, συντελεστές και άρα δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ αυτών των προστασιών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, ομοιομορφή ρύθμιση όσον αφορά την προσωρινή αποθήκευση των εμπορευμάτων και των αγαθών και όλα αυτά θα πρέπει βοηθήσουν στην ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος της μεταρρύθμισης του τελωνιακού κώδικα ήταν το να απλουστευτεί η διαδικασία τελωνισμού και να εξυγχρονιστεί η διαδικασία και να γίνει πιο εύκολη για τις επιχειρήσεις και να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια ηλεκτρονική διαδικασία. Ήταν μια πολύ καλή φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια πολύ καλή προσπάθεια την οποία εμείς ως Κοινοβούλιο χαιρετίζουμε. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία απειλούν ε, να ε, βγουν αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένα μιλώ για, το μη για τη μη προτιμησιακή καταγωγή. Εδώ μπορεί να υπάρχουν συνέπειες για μεγάλο τμήμα των, της διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, τρίτων χωρών και εδώ δίνει τη δυνατότητα πράξεων κατεξουσιοδότηση, ε, κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μακροχρόνιες διαδικασίες και θέματα τα οποία ήδη έχουν θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πιστεύω ότι δεν είναι ε, εφικτό να γίνει στην πράξη και δεν μπορούμε να έχουμε ε, ε, κανόνες και καταστάσεις απαριθμώντας διάφορες καταστάσεις το συζητήσαμε με την κυρία Λεγκρίπ και είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια διαφορετική αντιμετώπιση στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο καταλήγουμε σε μια συμβαστική λύση που δεν ξέρω κατά πόσο ε, θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι το εφικτό για να μπορέσει να προωθήσει ε, τους στόχους που είχε αρχικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι στο οποίο εμείς μπορούμε ως ομάδα να συμφωνήσουμε και ελπίζω ότι σύντομα και στην πράξη θα μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά για να μπορέσει το τελωνίο να λειτουργήσει καλύτερα και με μεγαλύτερη διευκόλυνση. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε από τους προηγούμενους συναδέλφους, φτάνουμε σε μια κατουσία θετική λύση μετά από μια μάλλον δύσκολη πορεία. Είναι δυνατόν να καταλήξουμε κάπου κάπου στην εργασία της ε, εισηγήτριας και των όσων συνεργάστηκαν μαζί της από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αυτός ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας, να διατηρηθεί όμως η προηγούμενη ασφάλεια, η προπάρχουσα ασφάλεια. Πιστεύω ότι στο τέλος, όπως είπε προηγουμένως η Εύελιν Γκέπαρτ, είναι σημαντικό η μη προσημειωτική ε, προέλευση να παραμείνει στον ορισμό όπως αναφέρεται στις συνθήκες. Θα ήθελα όμως να θεωρήσω ότι αυτό είναι ένα σημείο περάσματος και όχι η κατάληξη μιας διαδικασίας που θα πρέπει να έχει ως συγκεκριμένο στόχο τη μεγαλύτερη ενεχνευσιμότητα οποιοδήποτε προϊόντος Τέλος, το τελευταίο σημείο που θα θέλω να αναφέρω, κύριε Επίτροπε, είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την, την εποπτεία και τον έλεγχο από πλευρά της Επιτροπής. Γιατί μόνο μέσα από το, μια ενιαία συμπεριφορά και μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, πόροι ε, που δεν μπορούν εύκολα να νυχτευτούν, μπορούμε να έχουμε ένα τελωνιακό σύστημα που λειτουργεί σε επίπεδο τελειότητας. Εμείς ε, έχουμε δώσει στα τελωνία σημαντική Όπω αρμοδιότητες. Όπως γνωρίζετε αυτές αφορούν τον έλεγχο της πνευματικής ε, ε, ε, διοκτησίας, καταπολέμηση της απάτης κτλ. Όλα αυτά όμως θα μπορέσουν να επιτευχθούν εάν όταν προκύψουν προβλήματα που δεν μπορούν εύκολα να προβλεφθούν ή να προγραμματιστούν θα επιβληθούν οι απαραίτητες κυρώσεις. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που υπάρχει παραβίαση των κανόνων ή να υπάρχουν οι υπάρχοντες ε, οι απαραίτητοι πόροι. Συνεπώς, στην ουσία, ο ρόλος σας θα έλεγε αρχίζει ακριβώς εδώ. Γιατί το νομοθέτημα αυτό θα πρέπει να έχει μία όσο γίνεται μεγαλύτερη επίπτωση ξεκινάμε στην διαδικασία Catch the Eye και θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στη συνάδελφο Κόμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και την συνάδελφο εισηγήτρια γιατί εγώ είμαι υπέρ αυτού του νοσιακού κώδικα που προτάθηκε από την Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στη συνθήκη της Λισαβόνας καθώς και στους, ε, στις που έχουν επέρθει η ενιαία εφαρμογή αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να προκύψει όφελος για όλη την αγορά. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες μέσω της τεχνολογίας για να υπάρξει ένα περισσότερο δυναμικό περιβάλλον σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες αλλαγές που θα βελτιώσουν τον κώδικα. Για παράδειγμα την αξιοποίηση της, του κεκριμένου οικονομικού φορέα και την ε, ανάγκη για να υπάρχει μια δήλωση ε, με όχι, όχι κατεξουσιοδότηση πράξης. Και θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την εισηγήτρια. Eh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πραγματικά σύγχρονη νομοθεσία αυτή η οποία προκύπτει τώρα μετά την αναθεώρηση του ελληνικού κώδικα και νομίζω ότι έτσι θα ολοκληρωθεί η νέα αγορά. Έτσι θα έχουμε επίση ένα νέο σύστημα πληροφόρηση και πληροφοριών το οποίο ηλεκτρονικά θα μα βοηθήσει και θα μπορούν έτσι επιχειρήσει να μπορούν να επικοινωνήσουν από την έδρα του και θα μπορούν επίση να έχουν καλύτερη επαφή με τι τρονικές αρχέ και σε άλλο καλύτερο μέλο. Και επίσης αυτόν τον τρόπο θα μπορούν καλύτερα όλοι οι συναλλασσόμενοι να συμμορφωθούν με την τελωνική νομοθεσία και αυτό θα είναι καλό για τη διοίκηση των εμπορευμάτων, αλλά επίση ε, θα ωφεληθούν από αυτή την νομοθεσία και τελωνικέ αρχέ όσον αφορά την ανείχνευση του κάποιων ε, υπόπτων συναλλαγών, επιμάχων εμπορευμάτων και επομένω τώρα κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε ε, κάποια χρονικά πλαίσια για το πώς θα ε, δρούν όλοι τώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για τις ΜΜΕ. Ο κύριος Χάρμπορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πρόεδρος της Επιτροπής της Αρμοδίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κωνσταντς Λεγκρίπ και όλους τους κοιόδους ηγητές αλλά και συγητές που συνεργάστηκαν μαζί της και ξέρετε δεν ξέρω αν μας ακούνε οι συνεργάτες μας της Επιτροπής αλλά κατέβαλαν ε, Ηράκλειε προσπάθειε για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το κείμενο. Επίση, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ιρλανδική Προεδρία και α μην είναι εδώ, γιατί δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε το έργο μα χωρί τι προσπάθειέ του, κυρίω όσον αφορά τι εφαρμοστικέ πράξει. Και όπως είπε και η κυρία Γκέμπχαρτ, ε, τώρα δεν είναι τα θέματα τεχνικά, είναι πολιτικά. Οπότε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε εσάς αλλά και τους συνεργάτες σας για τη συνεργασία διότι νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικά τόσα κάνατε και έτσι όπως θα συμφωνείτε καταλήξαμε σε ένα καλύτερο νομοθέτημα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οπότε ε, έγινε αυτή η ζήτηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο από το 2006 ξεκίνησε σαν διαδρομή που κάναμε την κυρία Γκέμπχαρτ. Οπότε δεν μπορούμε τώρα παρά να έχουμε την εφαρμογή του νέου του ελληνικού κώδικα και ότι έχουμε σε αυτή τη νέα οδηγία ε, τα οποία τώρα θα τα προσέχει το κοινοβούλιο και θα πρέπει και τα κρατήμελη επίσης να μπορούν όλα αυτά να τα εφαρμόζουν. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για την λειτουργία της σωστικής αγοράς, είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους πολίτες, για τους αναλωσσομένους, όπως πάρα πολύ ορθά ενετόπισε η κυρία Μοσκαρντίνη. Έχουμε ζητήματα σε σχέση με παραποιήσεις, απομιμήσεις, με την ασφάλεια και επομένως τώρα τα τελωνία μπορούν να φροντίζουν το συμφέρον των πολιτών και τελικά αυτή είναι η δική μας αποστολή της δικής μας επιτροπής. Άρα σε όλους ε, ευχαριστίες και προσδοκώ αύριο ε, να γίνει ομόφωνη έγκριση της ε, Επιτροπής αυτής. Επιτροπή κύριε Σέμετα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον στο Κοινοβούλιο μας καταδεικνύει πόσο σημαντική υπόθεση είναι αυτός ο κώδικας για τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία ανέκαθεν πρόκειτο για κάτι πολύ σημαντικό, το εφαρμοστικό μέτρο και έχουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση στην Τελωνιακή Ένωση, κάτι το οποίο σημαντοδότησε την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθεσίας και ήταν το πρώτο βασικό βήμα, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας ενώπιση του 2020, να έχουμε αποδετική ε, ένωση, ένωση τελωνιακή και να έχουμε Υπηρεσίε υψηλή ποιότητα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό ο νέος ελληνικό κώδικα θα επιτρέψει στις τελωνικές αρχές να βελτιώσουν τι υπηρεσίε, θα μπορούμε να έχουμε καλύτερε υπηρεσίε προς τους αξιόπιστους συνεργασομένους και θα ωφεληθούν έτσι και οι Ευρωπαίοι πολίτε για όλε τι ενδυνάμει απειλέ, οπότε μπορούμε τώρα να στηριχτούμε στα ταχυδρομεία, να συνεχίσουν ε, το διακριτικό αλλά σημαντικό τους έργο με έναν τρόπο πολύ αποτελεσματικό για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Μάλκολμ Χάρμπορ για το έργο το οποίο επετέλεσε την κυρία Λεχρύπ ε, και τους σιώδες ηγητές. Όλοι ε, εργάστηκαν πάρα πολύ αξιόλογα ε, για ένα θέμα άκρος τεχνικό, τεχνοκρατικό, πολύ σημαντικό, οπότε και έτσι μπορέσαμε ε, να βρούμε κάποιους συμβασμούς για ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο και η Ελληνική Ένωση. Εγώ σε ευχαριστώ για τα γενικά σας λόγια και μας τους αδέλφους σας ευχαριστώ λέει πρόεδρος και τώρα να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Λουγκρίπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που έλαβαν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η ποιότητα των συζητήσεών μας ε, και η πυκνότητα ε, των θεμάτων που συζητήθηκαν δείχνουν ε, το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ενίσχυση της τελωνιακής διαδικασίας και για την βελτίωση των τελωνιακών διαδικασιών μέσα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Γνωρίζουμε ότι ακριβώς εκεί βρίσκεται ένα από τα κλειδιά της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πολλοί από τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο τόνισαν ότι χρειάζεται ένα ενιαίο σύστημα για τα 28 κράτη-μέλη. Ε, ήδη το έχουμε συζητήσει και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε προς μια λειτουργία πανευρωπαϊκή όσο δυνατόν αυτού του συστήματος των τελωνίων η απλούστευση, η βελτίωση των τελωνιακών διαδικασιών, η ελάφρυνση των, ε, του διοικητικού άχθους. Αυτή είναι η πορεία που θα μας οδηγήσει στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το στόχο από τα μάτια μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όπως ήδη είπαν αρκετοί ομιλητές, αυτά τα θέματα, τα τελωνιακά θέματα μπορεί να μοιάζουν ε, πεζά, τεχνικά, τεχνοκρατικά, ε, άνοστα. Στην πραγματικότητα όμως, μετά από 18 μήνες στο Κοινοβούλιο, ε, βλέπω ότι τα τελωνιακά θέματα βρίσκονται στον πυρήνα των οικονομικών και βιομηχανικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον πυρήνα των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε τη σημασία που έχουν οι τελωνιακοί δασμοί και η εισπραξή τους, αλλά παράλληλα ε, ενδιαφέρουν και άμεσα τους καταναλωτές μας, τους πολίτες μας, τους παραγωγούς μας και η ασφάλεια όλης αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να ενισχυθεί μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε με την ε, ανταγωνιστικότητα που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει χαρακτηρίζει. Με τις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση και με ε, τις πράξεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Μάρκον Χάρμπορ γενικότερα ε, μας περιμένει πολλή δουλειά τους επόμενους μήνες και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί την επιτήρηση που απαιτείται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ η ψηφοφορία για την έκθεση της συναδέλφου θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Η συνεδρίασή μας ε, ολοκληρώθηκε και οι εργασίες θα επαναληφθούν αύριο στις 9 το πρωί. Καλό σας βράδυ.